Οκ, Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ όλους αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν επεξηγήσεις ψήφου να φύγουν από την αίθουσα και μπορείτε να συζητήσετε έξω. Προχωρούμε λοιπόν στη διαδικασία επεξηγήσεων ψήφου. έκθεση Γκαβριέλ Μπάτο, πολιτές ε, σχέδιο ανάκαμψη για τον ερυθρό τόνο. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπιλμπά Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριο Μάτο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τον ερυθρό τόνο και για περιοχές όπως είναι τα Κανάρια. Τονίστηκε ότι πρέπει να είναι πιο δίκαιες οι ποσοστώσεις και πρέπει να λάβουν υπόψη τα κάτι μέλη τα σκάφη που ασκούν ε, βιοτεχνική και παραδοσιακή αλία που είναι πιο βιώσιμη. Αυτό ισχύει για τα Κανάρια. Το σχέδιο ανάκαμψης για τον τόνο έχει λειτουργήσει. Επομένως υπάρχει δυνατότητα να αυξηθούν σημαντικά <clears throat> οι ποσοστώσεις και αυτή η αύξηση των ποσοστώσεων θα πρέπει να αφορά τους παραδοσιακούς στόλους. <clears throat> Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω ότι ένας στόχο, στόλος βιοτεχνικής αλίας όπως αυτός των κανε, Καναρίων νησιών μπορεί μέσα σε 24 ώρες να καλύψει την ποσόστοση ενός μηνός. Γι' αυτό εγώ θέλω να πω ναι στην πρόταση αυτή για μια βιώσιμη αλία και μια πιο δίκαια κατανομή για τις ε, άδειες αλίας τόνου. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι έδωσα το λόγο στην κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Κανονικά οι κυρίες πρέπει να προηγούνται. <clears throat> Τώρα λοιπόν έχει το λόγο η κυρία Μπιλμπάο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτόν τον κανονισμό <clears throat> ο οποίος μεταφέρει τις ε, συστάσεις της ΙΚΑΤ και τις υλοποιεί σε ευρωπαϊκό δίκαιο, ακολουθώντας τις εμπειρογνωμοσύνες των επιστημόνων για να μπορέσει να ανακάμψει ο ερυθρό τόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ευαίσθητο οικοσύστημα τη Μεσογείου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά στον κόσμο. Επίση, όμω, είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η παραδοσιακή αλληλεία τόνου. Εδώ τίθενται ορισμένα σημαντικά θέματα. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα να υπάρξει ιδιαίτερη αναγνώριση στον παραδοσιακό τρόπο αλληλεία του τόνου με τράτες και άλλα παραδοσιακά σχήματα. Επίση πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη των θαλασσίων οικοσυστημάτων και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και την απασχόληση στον τομέα τη αλληλεία. Επίση, να εξασφαλίσουμε μια πιο ισοδίκια κατανομή των ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων και με ιδιαίτερο με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοτεχνική αλληλεία μικρή κλίμακο. Και τέλο, πρέπει να τονίσουμε τι αρμοδιότητε που πρέπει να διατηρήσει το Κοινοβούλιο στη μεταφορά των ε, συστάσεων των περιφερειακών οργανώσεων αλίας. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και δεν πρέπει να αποφεύγει το Συμβούλιο κάτι τέτοιο με ε, κατεξουσιοδότηση πράξη της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Παλώμα Λόπεθ Βερμέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρησιμοποιώ την ευκαιρία αυτή για να εξηγήσω γιατί κράτησα θέση αποχής για την έκθεση αυτή. Γιατί με τον κανονισμό αυτό, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάτι έχουμε χάσει. Και αυτό είναι τις επιπλέον ποσοστώσεις όσον αφορά τον, τον αυτό. Γιατί δεν ε, γίνεται μνήα στα μέσα τα οποία εμείς θέλουμε. Ο τόνος αυτός είναι τόνος ο οποίος αλλιεύεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο και προστατεύει πάρα πολύ την ε, οικολογική αλία, εκείνο ο οποίο με κυκλωτικά δίκτυα λέβεται. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι που γνωρίζει το σώμα και που πρέπει να υποστηρίξει πιο επίμονα απέναντι στις κυβερνήσεις του Συμβουλίου στο μέλλον. Εμείς δεν θα καταλήξουμε, δεν θα καταλήξουμε τη δικιά μας δέσμευση. Εμείς παρουσιάσαμε στην Επιτροπή Αλίας δύο πειραματικά προγράμματα με τα οποία προστατεύουμε την παραγωγή του τόνου με αυτόν τον τρόπο. Με μια ειδική σήμανση για αυτό το προϊόν. Είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι μπορεί να υπερψηφιστεί. Ευχαριστούμε. Τώρα, συνεχίζουμε. Δεν θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάτο, γιατί ο κύριος Μάτο ήδη μίλησε. Η κυρία Τζουφρίντα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση, διότι είναι καλό το πρόγραμμα του ΙΚΑΤ, ήταν επιτυχές και σήμερα οι θάλασσές μας και ιδιαίτερα η Μεσόγειος ε, είναι γεμάτες από ερυθρό Ρώσο. Όμως πρέπει να πω ότι έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να σεβαστούν τα όρια που επιβλήθηκαν και ακριβώς αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν και να ε, ψαρέψουν. Όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αύξηση των ποσοστώσεων μετά από την ανάκτηση του πόρου δεν ωφελεί σε τίποτα τους ψαράδες ομάδες. Οι μεγάλοι εφοπλιστές είναι αυτοί που εποφολούνται από την πλούσια σε τόνο θάλασσα και άρα ε, αυτό γίνεται εις βάρος χιλιάδων μικρών αλλιών και μικρών ε, επιχειρήσεων οικογενειακών που ζουν από την θάλασσα. Πρέπει με αυτούς να συνταχθούμε και να υποστηρίξουμε τα αιτήματά τους. Εγώ στηρίζω τη βιοτεχνική και μικρή, μικρής κλίμακας αλληλείας, τους ψαράδες που για αιώνες βασίζονταν ε, στη θάλασσα και τώρα διώχνονται από κανόνες και από οικονομικά συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με την την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Τζουφρίντα. Και τώρα έχουμε επεξήγηση ψήφου για την έκθεση του κύριου Ζαν Μαρή Καβαντά για τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση καθώς και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών ε, στοιχείων το, για τα διάφορα γαμικά καθεστώτα. Τζουφρίντα και πάλι. Σας ευχαριστώ. Υπερψήφισα αυτό το έκθεση γιατί η πραγματικότητα τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τους κανόνες και τις διατάξεις που πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα ενώπιον των προκλήσεων και των νέων ισορροπιών στην κοινωνία. Το Σέγγεν, το Έρασμος, η κινητικότητα ανάμεσα στα κράτη βοήθησαν τη γέννηση και τη διάδοση όλο ένα και πιο πολυάριθμων ευρωπαϊκών ζευγαριών ε, οικογενειών που ζουν σε κάποιο κράτος μέλος, έχουν σπίτι σε άλλο, ε, κληρονομούν ε, περιουσιακά στοιχεία σε ένα τρίτο κράτος μέλος. Είναι μια... Και ευτυχώς είχαμε τη δυνατότητα να ε, ε, ε, μάλλον είναι ζευγάρια που είχαν το θάρρος να περάσουν τα σύνορα και γι' αυτό και πρέπει και οι ευρωπαϊκοί κανόνες να προσαρμοστούν. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει τα κρατημέλη για να δώσει βεβαιότητα στα ζευγάρια και για να είναι σαφές το ποιος είναι ο αρμόδιος δικαστής κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είναι η μόνη περίπτωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ένα βουλευτή μπορεί να πάρει δύο φορέ συνέχεια το λόγο. Και περνάμε τώρα στην έκθεση. του κύριου Καβαντά όσον αφορά τις καταχωρισμένες σχέσεις. Ε, κύριος Πόσπισίλ. Είστε εδώ, μάλιστα. Παρακαλώ. Δεν πρόλαβα να πω ότι είναι θετικό το γεγονό ότι εγκρίθηκε αυτό ο κανονισμό. και θα ήθελα να θυμίσω μετά από τη συζήτηση που δίρκησε πάνω από πέντε χρόνια το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επιτέλου ενέκριναν ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι και τόσο δαφιλόδοξο γιατί αφορά μόνο κάποιου ε, επιμαχου ε, κανόνε και διατάξει ε, το πρόβλημα είναι ότι μόνο 18 χώρες μέλη ενέκριναν αυτό το σχέδιο και αυτό είναι προειδοποίηση και για το μέλλον καθώς ε, εάν δεν ε, παρέμβουμε, αν δεν κάνουμε κάτι για τα πιο επίμαχα άρθρα που αφορούν ας πούμε τις αρμόδιες δικαιοδοσίες ε, δεν, θα δεν μπορούμε εκεί να βρούμε συμφωνία. Είναι καλό το σχέδιο, αλλά όπως είπα μόνο 18 χώρες το ενέκριναν, άρα αποδυναμώνεται. Γιατί μόνο σε ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ισχύει. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτό μας λυπεί. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Πόσπισιλ. Και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου για το ψήφισμα ε, που αφορά τις σφαγές στο Ανατολικό Κονγκό. Το λόγο έχει η κυρία Τζουφρίντα. Εγώ υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, διότι είναι δίκαιο από τις Βρυξέλλες να ακουστεί η κραυγή ε, της ε, Φρίκης και να εγκριθεί ένα ψήφισμα από τις Βρυξέλλες για το τι συμβαίνει εκεί. Δεκάδες δολοφονίες παιδιών και γυναικών εδώ και χρόνια στο Ανατολικό Κονγκό γίνονται δολοφονίες και σφαγές ε, ενώ ευημερεί το καθεστώς το οποίο γυρνά τα μάτια, στρέφει τα μάτια του άλλου. Ασχολούνται με πολύ πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις ε, που αναγκάζουν ας πούμε πάνω από 35.000 οικογένειες να φύγουν από τα σπίτια του δεν μπόρεσαν να σταματήσουν εκεί τις σφαγές ε, που είναι πολύ ανησυχητικές εκτός που προκαλούνται αδίκως θύματα ανάμεσα στον ε, άμαχο πληθυσμό ε, βαραίνει στη συνείδηση του ΟΗΕ και τη διεθνούς κοινότητας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο ισχυροί. Κανένα κόμπακτ για τη μετανάστευση δεν μπορεί να, είναι, να λειτουργήσει εάν δεν επικρατήσει ειρήνη στην Αφρική. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Κέγγε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καμία ε, συγχώρεση για όσους κάνουν τέτοιες σφαγές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφωστά εκφράστηκε για τις σφαγές που καταστρέφουν ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη περιφέρεια στο Ανατολικό Κονγκό. Έχει Έχουμε ε, ε, ε, παρέμβει μόνο περιστασιακά. Εάν δεν σταματήσει αυτή η κατάσταση, μπορεί να οδηγήσει σε γενοκτονία που θα αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Το καθεστώς που σοβεί και έχει ένα χαρακτηριστικό ε, για τους λαούς που κατοικεί ε, σε αυτές τις περιοχές. Ε, δεν θα, θα αισθανόμαστε ντροπή και είμαστε με τους λαούς Μπένι, Μπουτέμπο και Μπουτέρο. Ευχαριστώ κυρία Κέγγε. Και τώρα περνάμε στην έκθεση σε αιτιολογικέ μάλλον ε, σε τη ψήφου σε σχέση με την έκθεση του κ. Κράσνοντεύσκη για την υλοποίηση στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο τομέα τη εκπαίδευση και της κατάρτισης. Κυρία Τζουφρίντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω ε, κάθετα ότι τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μεγάλο τμήμα αυτών των δυσκολίων που αντιμετωπίζει, μπορούν να ε, ξεπεραστούν μέσω της παιδείας και της κατάρτιση. ριζοσπαστική η ε, ριζοσπαστικοποίηση, ο θρησκευτικό τα κτλ. μπορούν να ξεπεραστούν μέσω μια ε, σωστή παιδεία, μέσα από τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα πολιτιστικά κέντρα κτλ. Και δεν είναι μόνο τα σχολεία και εκπαιδευτική. Η κατάρτιση είναι και άτυπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το διαβατήριο των δεξιοτήτων ώστε να δώσει όλο ένα και περισσότερη αξία στι δραστηριότητε εθελοντισμού και συνεργασίας ε, σε ΜΚΟ. Ειδικά ε, για όσους δεν θέλουν να βαθύνουν στις, μελέ, στις σπουδές, η διαδικασία, ε, θελοντική διαδικασία αναγνωρίζεται ε, και θα πρέπει να στηρίξουμε τον πολιτισμό, την παιδεία και την κατάρτιση για να δώσουμε στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες να οριμάσουν ως Ευρωπαίοι πολίτες και ως επαγγελματίες που μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα τους υπολείπους. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την επεξήγηση ψήφου και τώρα έχουμε τις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση της κυρίας Παλώμα Λόπες Βερμέχο, ανανεώσιμη ενέργεια και σχετική έκθεση πρόοδου και δίνω το λόγο στην κυρία Τζουφρίντα. Εγώ υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί είμαι βεβαία ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι το μέλλον για την Ευρώπη και όχι μόνο λόγω τη περιβαλλοντική του αλλά και για να δώσουν όθηση στι διάφορε περιφέρειε, περιφέρειε όπω η δική μου, η Σικελία, στην Νότια Ιταλία και στην Νότια Ευρώπη, που θα μπορούσαν να λειτουργήσει ω ε, πειραματικό τόπο για την ανάπτυξη των, των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια ε, και να είναι και μάλιστα αυτόνομη ε, και όχι επίπεδα ρήπανση ε, φοβερά και τρομερά και ακόμα γίνεται λόγο και για πετρέλαιο. Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση, αλλά πρέπει να βοηθηθούν και οι περιφέρειε για τη δαπάνη των διαφθορτικών ταμείων, γιατί στην ε, ε, πολιτική συνοχή στο ποσοστό που πάει στην ανανεώσιμη ενέργεια είναι 1,4% μόνο. Και πρέπει επίση να δρομολογηθούν οι πόροι που απευθύνονται στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια προ τι περιφέρειε που είναι πλούσιε από πόρου, αλλά είναι πιο αδύναμε όσον αφορά τον σχεδιασμό. Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι το κλειδί για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία πιο καθαρών πόλεων, πιο υγιούς περιβάλλοντος και μια καλύ... μιας καλύτερης Ευχαριστώ και την κυρία Τζουφρίντα. Και τώρα τον λόγο έχει η κυρία Μπιλιάνα Μπόρζεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονό ότι η Κροατία είναι μεταξύ των χωρών αυτών που είναι πολύ κοντά στο να επιτύχουν του στόχου που έχει θεσπίσει η Κομισιόν. Θέλω να υπογραμμίσω και τη σημασία τη καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή <clears throat> και σε ό,τι αφορά το ρόλο του ω δυνητικών παραγωγών ενέργεια. Οι καταναλωτέ θα πρέπει να μπορούν να έχουν μια σαφή ανάγνωση τη κατανάλωση ενέργειά του για να μπορούν να την ελέγχουν. Μπορεί ένα νοικοκυριό να, σώσει, να εξοικονομήσει μέχρι 30% ενέργειας στην ψήξη και, στην, και στη θέρμανση. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή τη νέα πρωτοβουλία για να απλοποιηθούν οι διάφορες κατηγορίες ενέργειας για τους καταναλωτές και η Επιτροπή Ενέργειας έχει δεχτεί μια πρόταση της ομάδας των σοσιαλιστών για την ε, δοκιμασία των συσκευών όχι μόνο σε εργαστηριακές αλλά σε πραγματικές συνδίκες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι μελέτες οι οποίες αφορούν για τα σφάλματα των μηχανισμών αυτών πρέπει να συζητηθούν. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανανεώσιμη <clears throat> ενέργεια και να δώσουμε περισσότερη επιλογή στους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί. Συγχαρητήρια για την ε, κροατική ποδοσφαιρική ομάδα, λέει ο πρόεδρος έδειξαν ανανεώσιμη ενέργεια στη νίκη τους κατά της Ισπανίας. Και τώρα ο κύριος Σόγκορ, τον οποίο θέλω να συγχαρώ επίσης, γιατί και η Ουγγαρία τα πάει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Σόγκορ. Ο κύριος Σόγκορ είναι, είναι απόνομος από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Σον Κέλλη έχει το λόγο. Τελευταίος αλλοχίστατος. ευχαριστώ. Και εγώ με μεγάλη χαρά έχω υποστηρίξει την έκθεση αυτή, όπως και οι περισσότεροι βουλευτές της ομάδας μας. 444, όπως ξέρετε, ψήφισαν υπέρ και μόνο 133 κατά. Όλο αυτό μας καταδεικνύει ότι τα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που διατυπώθηκαν στην COP21 στο Παρίσι. Και τώρα έχουμε μια θαμάσια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια. Όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, στην αρχή της εντολής του θα πρέπει να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, ένα ηγετικό ρόλο στα θέματα αυτά και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα μέσα από την έρευνα. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια γίνεται και έρευνα για την θαλάσσια των κυμάτων και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε τέτοιες τεχνολογίες πρέπει να τι χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο Κύριε Κέλλη. Και τώρα περνάμε στην λουκούμια έκθεση του κυρίου Πίπα, έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Και εδώ έχουμε πρώτα την κυρία Τζουφρίντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση για την ε, ενεργειακή απόδοση και επάρκεια, γιατί είναι πολύ κρίσιμο θέμα για το προβληματισμό μας και για τον ορισμό νέων στόχων για το περιβάλλον, για την ενέργεια και το κλίμα. Ήταν η χρονιά της COP21 που όρισε ε, ε, φιλόδοξους στόχους για ένα περιβάλλον το οποίο σίγουρα υποφέρει. Και έπειτα η Ευρώπη ε, ε, δεν είναι, είναι σε θέση ε, μάλλον αμφισβητείτε αν θα μπορέσει να επιτύχει το στόχο της μείωσης του 20% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, συγκρούονται η δημοκρατία με την οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα πρέπει η Ευρώπη να τα, να, να τα αντιμετωπίσει αυτά. Οι ενεργειακοί στόχοι, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και ένα σωρό άλλοι για να είναι αποτελεσματικοί δεν μπορούν παρά να είναι α, ε, προσαρμόσιμη στις οικονομικές αλλαγές, στις οικονομικές κρίσεις, ε, για να, στόχο που θεωρεί να έχουμε την πράσινη οικονομία ε, για να μπορέσει να ανακάμψει και ολόκληρη η οικονομία. Ευχαριστώ κυρία Τζουφρίντα. Ε, Ευχαριστώ την κυρία Τζουφρίντα. Τώρα ο κύριος Σον Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πάλι. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική έκθεση και υπήρξε αμφιλεγόμενη. Πρέπει όμως να επενέσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Πίπα, ο οποίος είναι από τη δική μου ομάδα και ο οποίος έκανε, έκανε πολύ καλή δουλειά και κατάφερε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμβαστικές λύσεις. Γι' αυτό καταφέραμε να έχουμε μια σειρά από σημαντικές ψηφοφορίες που ευδοκίμησαν και εμείς έχουμε τονίσει ως ομάδα μας ότι ε, είπαν ορισμένοι ότι πρέπει να καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση, αλλά εγώ δεν ακολούθησα τη θέση της ε, ομάδας μου. Ήμουνα, σκέφτηκα τη δική μου χώρα, ήμουνα και εγώ στο Παριστίν COP21, είδα πόσο σημαντική είναι η <clears throat> ανανεώσιμη ενέργεια και γι' αυτό η, μάλλον η αποδοτικότητα της ενέργειας και γι' αυτό υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Ελπίζω να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη διαμάχη. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Κύριε Κέλλη, μπορείτε να είστε υπόδειγμα για μένα σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρόνου αγόρευσης σε επεξηγήσεις ψήφου. Συγχαρητήρια λοιπόν. Και ο τελευταίος ο, ομιλητής είναι ο κύριος ε, Κόρβιν Μίκε. Βέβαια η βίβλος λέει «Οι ίστατοι έσονται πρώτοι». Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος θα λάβει το λόγο από τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Κόρβιν Μίκε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς καταψηφίσαμε και τις δύο εκθέσεις για την ενέργεια. Επομένως είμαι εξοργισμένος για το γεγονός ότι κάποιοι αναλφάβητοι και ανεγκέφαλοι μιλούν για θέματα τα οποία αγνοούν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρώπη δεν προχωρά. Η Ευρώπη μένει πίσω. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε όταν το φυσικό αέριο είναι τέσσερις φορές φτηνότερο από ό,τι στην Ευρώπη και είναι τρεις φορές φθηνότερο στην Κίνα. Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όχι μονάχα θα πρέπει να καταληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιστεύω ότι αυτή οι οποίοι προπαγανδίζουν υπέρ της κλιματικής αλλαγής και θέλουν να καταστρέψουν τις ευρωπαϊκές ενεργειακές ε, πηγές θα πρέπει να συρθούν ενώπιον του δικαστηρίου και να καταδικαστούν για αυτά που έκαναν στην ανθυρή περιοχή της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Κόρβιν Μίκε. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν τη διαδικασία εξήγησεων επεξηγήσεων ψήφου. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ το προσωπικό και τους διερμηνείς. Καλό μεσημέρι και τα πρακτικά της συνεδρίας αυτής θα διαβιβαστούν στο Κοινοβούλιο στην